νέοι να μπορούν να σπουδάσουν όπως πρέπει, να αποκτήσουν προσόντα και να δουλέψουν εκεί που θέλουν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Τελειώσαμε με αυτή την παρέμβαση, ε, τη συζήτηση αυτή. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση HARMS για τη χρηματοδοτική συνδρομή της κοινότητας για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοσλόντουι στη Βουλγαρία. Μιλάμε για το πρόγραμμα Κοσλόντουι. Κυρία Χάρμς, έχει τέσσερα λεπτά για να ξεκινήσει η συζήτηση. Η κυρία Χάρμς, λοιπόν, η συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αρκετά γενναιόδωρος ο χρόνος απόψε. Καταρχήν ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις με την Κομισιόν και με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη Βιομηχανική Επιτροπή και την Επιτροπή Ενέργειας. Δεν είμαστε πάντοτε σύμφωνοι, αλλά σε ένα συμφωνούμε, ότι δηλαδή χρειάζεται ευρωπαϊκή κοινή υποστήριξη για την Βουλγαρία κατά την αντιμετώπιση του κόστους του, της παύσης λειτουργίας των τεσσάρων μπλοκ στο Κοσλοντούι. Πρέπει να το τονίσω αυτό. Το 2006 340 εκατομμύρια έλαβε η Βουλγαρία, το 2007 μέχρι το 2008 253 εκατομμύρια ευρώ, το 2009 89,5 εκατομμύρια ε, διοχετεύθηκαν προς τη Βουλγαρία και αύριο στην ψηφοφορία θα αποφασίσουμε περαιτέρω συμβολές 300 εκατομμυρίων ευρώ από την Ένωση προς τη Βουλγαρία. Ω ένδειξη αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη γιατί η βουλγαρική κυβέρνηση στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι είναι έτοιμη ε, να δεχτεί τα προβλήματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων στο Κοσλοντούι και γι' αυτό θα πρέπει, συμφώνησε να κλείσει τους αντιδραστήρες. Με την έκθεσή μου προσπάθησα για το τελευταίο κομμάτι, την τελευταία δόση, τη... υποθέτω ότι θα είναι η τελευταία δόση, ε, προσπάθησα να επιτύχω μια αλλαγή, μια τροποποίηση. Θα ήθελα να προτείνω τα χρήματα τα οποία δεν είναι άμεσα για τον παροπλισμό, τον decommissioning και την ε, ε, διαχείριση των αποβλήτων για το ενδιάμεσο, την ενδιάμεση εγκατάσταση και το Κοσλοντούι ε, έχουμε μια υπέρβαση 120 εκατομμυρίων, τουλάχιστον μέρος αυτών των χρημάτων θα έπρεπε να επενδυθούν στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της τελικής αποθήκευσης ε, υψηλής ραδιενέργειας καταλήπων στη Βουλγαρία και να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα ταμείο που θα αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα τα οποία δεν ε, έχουν γίνει μέχρι τώρα στην Βουλγαρία. Μέχρι τώρα δεν κατάφερα να πείσω την πλειοψηφία στις επιτροπές ε, υπέρ αυτής της ιδέας. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία. Στις συμβιβαστικές τροπολογίες που διαπραγματευτήκαμε στις επιτροπές πάλι ε, προσπάθησα να διατηρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, σε σχέση με την ε, αποθήκευση, τελική αποθήκευση και η ενδιάμεση αποθήκευση εντάσσεται εδώ, θα ήθελα η Κομισιόν να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το συγκεκριμένο κόστος. Τι στοιχίζουν όλα αυτά στο Κόσλο πόσα, πόσα χρήματα χρειάζονται για το κλείσιμο και την ε, σωστή ε, επεξεργασία και αποθήκευση των ε, αποβλήτων. Δεύτερον, τα χρήματα που θα στείλουμε στη Βουλγαρία δεν θέλω να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στο, στον άνθρακα, ε, γιατί αυτό δεν αποκλείεται από ό,τι φαίνεται. Κατά τα άλλα, χαίρομαι διότι η έκθεση έδωσε το έναυσμα για μια ζωηρή πολιτική συζήτηση ε, σε σχέση με την αποθήκευση των ατομικών αποβλήτων γενικά. Ε, ήδη σχεδιάζεται η οδηγία και την περιμένω με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Εκ μέρους της Κομισιόν έχει το λόγο ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, υπάρχει στο, στην ημερήσια διάταξη απόψε ένα ενεργειακό θέμα, δηλαδή η παράταση της χρηματοδότησης προς τη Βουλγαρία για τον παροπλισμό στο Κοσλοντούι. Ένα θέμα ευαίσθητο, σημαντικό και γι' αυτό χαιρετίζω την επικοδομητική στάση σας. Ευχαριστώ για αυτήν. Το θέμα συζητήθηκε με την εισηγήτρια την κυρία Χάρμσε ε, και τις αρμόδιες επιτροπές. Συζητήθηκε ε, επί μακρόν. Η έκθεση της Κομισιόν ε, σε μεγάλο βαθμό συνάδει με τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ για την υποστήριξη σε σχέση με τα 300 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό σύμφωνα με το γενικότερο συμφέρον της Ένωσης και χάρη της ασφάλειας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Δεύτερον, η έμφαση στην περαιτέρω βοήθεια θα πρέπει να στοχεύει στον, στον παροπλισμό και γι' αυτό υπάρχει ε, ένα κατάλληλο ε, ε, ποσό των 180 εκατομμυρίων. Επίσης, υπήρξαν οικονομικά προβλήματα που εξηγούνται ιστορικά στην Βουλγαρία. Ε, πάντως, το σημαντικότερο είναι να υπάρξει ε, πλήρης χρηματοδότηση για τον παροπλισμό. Θα ήθελα να τονίσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ε, τροπολογιών μπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή. Για λόγους χρόνου δεν μπορώ να επισέλθω σε όλες. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τη θέση της Κομισιόν σε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Δύο θέματα που και στην έκθεση ε, αναφέρονται και μέσα από τροπολογίες και από την εισηγήτρια την κυρία Χάρμς. Μιλάω πρώτον για τη συνέχιση της οικονομικής υποστήριξης για μέτρα στον ενεργειακό τομέα εκτός από την επιθυμία της βουλγαρικής κυβέρνησης υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της οικονομικής ε, της χρηματοδότησης. Ε, μιλάμε για ίση μεταχείριση με την Λιθουανία και τη Σλοβακία όπου αντίστοιχα μέτρα προωθήθηκαν ε, και προβλέπονται μέχρι το 2013. Επίσης, ε, ε, μέτρα στον τομέα ενεργειακής απόδοσης. Τα εργοστάσια στη Βουλγαρία έχουν, που χρησιμοποιούν άνθρακα έχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, η, δυνατότητα, η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξε στη Βουλγαρία ε, με την ατομική ενέργεια. Ε, έτσι λοιπόν η Βουλγαρία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να υποστηριχθούν ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν ε, και στο μέλλον μέτρα στον ενεργειακό τομέα όπως και για την υποδομή του δικτύου. Δεύτερον, το θέμα υποστήριξη για την ανάπτυξη μιας ε, σωστής αποθήκευσης ε, των προϊόντων καύσης. Η Κομισιόν ε, συμφωνεί με την εισηγήτρια εις ό,τι αφορά την αναγκαιότητα μιας λύσης για την σωστή αποθήκευση των προϊόντων της καύσης. Στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος Κοσλοντούι όμως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, στον ε, πυρηνικό τομέα. Αν και η αποθήκευση των προϊόντων καύσης αποτελούν κομμάτι των ε, καταλήπων, ε, δεν δεν έχουν σημασία πέραν του κλεισίματος ε, των αντιδραστήρων. Είναι σημαντικό να ε, καλύψουμε τα ενδιάμεσα στάδια, πράγματα που ε, προβλέπονται ήδη. Η τελική αποθήκευση όμως δεν είναι το αποτέλεσμα του κλεισίματος των τεσσάρων μονάδων του Κοσλοντούι. Να υποστηρίξω ότι η Κομισιόν, όπως είπαμε ήδη, το θέμα της αποθήκευσης το ε, ε, βλέπει ε, με πληρότητα και επίσης θα υποβάλει πρόταση για την αποθήκευση ραδιενεργών υλικών και την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων καύσης. Υπολογίζω στην επικοδομητική σας υποστήριξη και προβλέπω ότι θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τέλος, συνοψίζω ως εξής. Η Κομισιόν χαιρετίζει το γεγονός ότι συμφωνεί το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν να ε, συνδράμει με 300 εκατομμύρια ευρώ τη Βουλγαρία την επόμενη τριετία. Ε, χαιρόμεθα διότι το, η έμφαση δίνεται στην ε, ασφάλεια σε ό,τι αφορά τα μέτρα και επίσης χαιρετίζομαι τα προγράμματα που θα υποστηριχθούν στον ενεργειακό τομέα γενικότερα. Η περαιτέρω χρηματοδότηση που υποστηρίζεται ε, είναι ένδειξη αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βουλγαρία και συμβάλλει σημαντικά στην πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης επίσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο λόγος για δύο λεπτά στην κυρία Παρβάνοβα. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, като докладчик в Комисията по околна среда бих искал... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς υπερψηφίσαμε σε επίπεδο επιτροπής αυτήν την έκθεση. Χαίρομαι που οι προτάσεις μας εντάχθηκαν στην έκθεση και το Κοινοβούλιο μπορεί πλέον να δώσει ένα σαφές μήνυμα για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον παροπλισμό και την αποξύλωση του σταθμού του Κοσλοντούι. Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει την, τον ασφαλή παροπλισμό σύμφωνα με, τα πιο υψηλά, σύμφωνα με τις πιο υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Θα, ένα τμήμα του, της χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για περιβαλλοντικούς σκοπούς και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπήρξαν, μάλλον ασκήθηκαν πιέσεις για πολιτικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους και είναι πολύ σημαντικό που εξασφαλίζουμε την κατάλληλη αποζημίωση της ε, Βουλγαρίας ε, για το κλείσιμο του σταθμού, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε ότι το παρελθισμό θα γίνει με ασφάλεια. Η ε, τελική απόθεση του πυρηνικού υλικού είναι πολύ σημαντική βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει μόνη τη Βουλγαρία. Είναι μια πρόκληση που απαιτεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική και ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κυρία Χάρμς, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι η Βουλγαρία δεν έχει επουδενή σκοπό να χρησιμοποιήσει αυτά τα, αυτό, αυτή τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία καινούριων ε, σταθμών παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα. Σκοπεύουμε να σεβαστούμε πλήρως την κοινοτική νομοθεσία και να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνολογία. Είμαστε υπεύθυνοι χώρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παρβάνοβα. Εποφελούμε τις ευκαιρίες για να σας πω, να σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο αργά. Γιατί η αγαπημένη μου οι διερμηνείς, οποίους ακούω στα ακουστικά μου, εκπέμπουν ε, σως κάθε τόσο όταν μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και αν μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν μεταφράζεστε, ε, καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που καταλαβαίνουν τη γλώσσα σας. Και δεν χρειάζεται να ακούν τη διερμηνία. Παρακαλώ λοιπόν να επιβραδύνετε λίγο. Ωραία. Ομιλητές εξ ονόματος ε, πολιτικών ομάδων. Καταρχήν ο κύριος Ουρούτσεφ για δύο λεπτά εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την πίεση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, η Βουλγαρία συμφώνησε να κλείσει τους τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες στο Κοσλόντουι και με βάση τους συμπεφωνημένους όρους το έκανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε οικονομική βοήθεια ε, στην περίοδο 2007-2009 για να βοηθήσει για τον παροπλισμό και κλείσιμο των μονάδων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε και εγγυήσει για τη συνέχιση της υποστήριξης για την περίοδο 2010-2013. Με αυτόν τον τρόπο με βάση τους όρους της οικονομικής ενίσχυσης, η Βουλγαρία θα παίξει ισότιμο με τη Σλοβακία και την Λετωνία, που επίσης προέβησαν σε πρόορη σε και παροπλισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Ε, στα πλαίσια της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτή την πρόταση. Το ποσό το επιπλέον που, δίνουν στη Βουλγαρία δεν μπορούν να την αποζημιώσουν για την απώλεια δισεκατομμυρίων από την πρόορη, λόγω της, της του πρόορου κλεισίματος και παροπλισμού του πυρηνικού εργοστασίου. Είναι πολύ σημαντικό ε, να εκμοντερνιστεί ο τομέας τη ενέργειας, να μειωθούν οι επιβλαβείς ε, εκπομπές, να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια και εξοικονόμηση της ενέργειας. Η έκθεση που ψηφίστηκε στην Ήτρε με μεγάλη πλειοψηφία ακριβώς αυτό θέλει να εξασφαλίσει. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε με τις ανανεωμένες απόπειρε να μπουν κάποια σχόλια ε, στο κείμενο για τις ε, εγκαταστάσεις που πυροδοτούνται με άνθρακα. Προτείνουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν και να απορρίψουμε τις νέες πέντε ε, τροπολογίες των πράσινων. αυτά, ευχαριστώ. Εκ μέρους του Σοσιαλιστικού, της Σοσιαλιστικής Ομάδας, ο κύριος Κάλφιν για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και, την εισηγήτρια και την Κομισιόν. Ιδιαίτερα τον κύριο Ότιγκερ για το έγγραφο το οποίο υπέβαλε. Κυρία Χάρμς, κατέβαλε πολλές προσπάθειες κατά τη συζήτηση του εγγράφου και έθιξε σημαντικά για τους ευρωπαίους πολίτες θέματα. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η Βουλγαρία στον παροπλισμό των ε, αντιδραστήρων του πυρηνικού της σταθμού Κοσλοντούι. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι, αλλά δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει αναλάβει αυτή την δέσμευση, θα πρέπει να την υλοποιήσει. Το κλείσιμο ενός τέτοιου μεγάλου πυρηνικού σταθμού νωρίτερα από, το προβλεπόμενο, από την προβλεπόμενη ημερομηνία α, συνεπάγεται πρόσθετα άμεσα και έμεσα κόστη που εν μέρει καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σημερινή πρόταση η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση στην Βουλγαρία με αυτήν που επεφύλαξε σε άλλες χώρες που ανέλαβαν παρόμοιες δεσμεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ε, πολιτική ευρωπαϊκή συνοχή. Το 60% των ε, κονδυλίων ε, θα προοριστούν άμεσα στην αποξήλωση. Το υπόλοιπο 40% προορίζεται για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για την μείωση των επομών διοξιδίου του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έθιξαν διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα, τι θα γίνει με, το, με τα ακτινοπολιμένα στοιχεία και το υπόλοιπο καύσιμο. Το έθιξε και ο κ. Σότιγκερ σήμερα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το φθινόπωρο ε, θα υποβάλει μια ιδιαίτερη οδηγία για αυτό το ζήτημα και το Κοινοβούλιο θα συζητήσει. Ε, λοιπόν, αυτή την οδηγία σε βάθος είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες μας ζήτημα. Συνεπώς, αυτή τη ε, στιγμή η αποσημείωση που δίνουμε στην ε, Βουλγαρία ε, η αντιστάθμιση αν θέλετε δεν προδικάζει την ε, θέση που θα λάβουμε το φθινόπωρο. Ε, αυτή η χρηματοδότηση δηλαδή δεν αποτελεί προηγούμενο και δεν θα πρέπει να νοηθεί ως τέτοια. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την ευθύνη των χωρών που διαθέτουν τέτοιου είδους αντιδραστήδες, την ευθύνη τους να βρουν μια, ένα ασφαλή τρόπο ε, απόθεσης των ε, εκτινοπολιμένων στοιχείων και του καυσίμου. Ε, επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κλείσιμο του Κοσλοντούι δεν θα αυξήσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα θέλαμε το κείμενο να καταδείξει την συνέπεια και την συνέχεια της κοινωτικής πολιτικής. Τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το λόγο τον οποίο χορηγούνται, με διαφάνεια. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, τα κονδύλια αυτά θα τροφοδοτήσουν ένα ειδικό ταμείο στο οποίο καταλήγουν δωρεές και άλλων χωρών. Ε, σύμφωνα με τους ε, κανόνες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν με βάση συγκεκριμένα προγράμματα και το ελεγκτικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ελέγξει τη χρήση τους. Ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Κάλφιν. Πρόεδρος. Ε, εκ μέρους των φιλελευθέρων, για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Βάλεαν. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε. Ως εισηγήτρια για τις ενεργειακές υποδομές, είμαι πολύ ευαίσθητη σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Είμαι Ρουμάνα και γι' αυτό ακριβώς ενδιαφέρομαι τα μάλα για αυτό το θέμα του πυρηνικού εργοστασίου του Κοσλόντουι. Είναι στα σύνορα με τη χώρα μου και γι' αυτό ακριβώς μας ανησυχούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους. Το εργοστάσιο Κοσλόντου είναι 4 χιλιόμετρα από τον ε, Δούναβη και 150 χιλιόμετρα από το Βουκουρέστι. Με βάση διεθνείς ε, πραγματογνωμοσύνες ε, δεν υπάρχει κάλυμα προστατευτικό και υπάρχει πρόβλημα ραδιενέργειας στον υδροφόρο ορίζοντα και μόλυνση στον τροφόρο ορίζοντα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την, τον παροπλισμό και θα πρέπει να δοθούν επαρκή κονδύλια σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να, να κρατήσουμε ψηλά τα πρότυπα τη ασφάλεια, να υπάρχει η πραγματική η πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται και να εφαρμοστούν οι διεθνεί καλύτερε πρακτικέ. Η αποξύλωση θα πρέπει να γίνει με βάση αυστηρού κανόνε και πρότυπα, αλλιώ θα δημιουργήσει κινδύνου ασφαλεία σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω πραγματικά αυτή την πρόταση και υποστηρίζω να δοθούν επιπλέον 300 εκατομμύρια σε αυτό το σκοπό. Ε, πριν από λίγους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίδοντας 75 ε, εκατομμύρια στα πλαίσια του προπολογισμού του 2010 έδειξε ε, μια ένα έντονο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει διαφάνεια για την χορήγηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της χρηματοδότησης ε, και του τρόπου που ξοδεύονται. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε ποιες είναι, ποια είναι τα θετικά σημεία και τα αρνητικά σημεία του προγράμματος, ούτω ώστε να δούμε την επόμενη περίοδο χρηματοδότηση 2010-2013 μαζί με τα, ε, τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης πώς πρέπει να ξοδευτούν αυτά τα κονδύλια. Ε, θα πρέπει η Βουλγαρία να παρουσιάσει την εθνική στρατηγική της θα πρέπει να μας μιλήσει για το πώς θα προωθήσει τα νεώσιμε ε, πηγές ενέργειας για να πάρει και τα, το, το ποσό των 120 εκατομμυρίων ε, ευρώ το ποσό αυτό που προβλέπετε. Κοιτάξτε. Κυρία Βαλέν, ε, το χρόνο σας κατά πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Στογιανόφ χρησιμοποιώντας ε, τον κανόνα της μπλε γαλάζιας κάρτας ζήτησε να σας κάνει μια ερώτηση. Μ' ακούτε κύριε Βαλέαν. Κύριε Βαλέν, σε εσά απευθύνομαι. Ο κύριο Στοιανόφ, ε, χρησιμοποιώντα τον κανόνα τη γαλάζια κάρτα, μου ζητάει να σα κάνει μια ερώτηση. Θα μπορούσατε να απαντήσετε. Κύριε Στοιανόφ, έχετε ένα λεπτό για να αποβάλλετε την ερώτησή σα. Ε, ναι, έχω μια πολύ συγκεκριμένη και σύντομη ερώτηση. Ε, η κυρία Βαλεάν ε, έκανε μια ερώτηση για την ασφάλεια. Πριν την αποξύλωση των τεσσάρων μικρότερων μονάδων του Κοσλοντούι, ε, αυτές είχαν αποκληθεί οι πιο ασφαλείς μονάδες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Κύριε Βαλέαν, έχει το λόγο. Uh, well, colleague, uh, chair, what can I... Αγαπητέ συνάδελφε, τι να απαντήσω. Έχουμε τρελαθεί όλοι μας. Ποιος ο λόγος ε, που λέγονται αυτά. Νομίζω ότι έτσι αποφασίστηκε από πολλούς ανθρώπους και εμείς θέλουμε να τους ακολουθήσουμε, να τους υποστηρίξουμε. Αλλά τι άλλα να σας πω. Ουδέν σχόλιον. Εξ τη της ομάδας των Πρασίνων, για ένα λεπτό ο λόγος του κύριο Τρεμόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στη σημερινή μας συζήτηση ότι την τελευταία δεκαετία η ευρωπαϊκή ένωση έδωσε στη βουλγαρία για το κλείσιμο των τεσσάρων μονάδων του κοζλοντούι 550 εκατομμύρια ευρώ. δίνει τώρα άλλα 300 εκατομμύρια σύνολο 850 εκατομμύρια χωρίς να υπολογίσουμε τα τεράστια ποσά τα οποία έχουν δοθεί για επιδιορθώσεις και αύξηση της ασφάλειάς του. δηλαδή το πυρηνικό αυτό συγκρότημα το έχουμε πληρώσει περίπου χρυσό και για κάποιους ήταν και χρυσοφόρα η ελλάδα. παρ' όλα αυτά η επιτροπή συνεχίζει την έμεση χρηματοδότηση του πυρηνικού λόμπι. εμείς ζητούμε να μην γίνουν άλλα παζάρια με τη βουλγαρική κυβέρνηση. το κοινοβούλιο μαζί με την επιτροπή να διασφαλίσουν την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και να τη θεωρήσουν μέρος του προγράμματος απόσυρσης. ως πράσινοι ζητάμε το υπόλοιπο 40% των 300 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος για την απόσυρση των πυρηνικών αντιδραστήρων να διοχετευθεί από τη βουλγαρική κυβέρνηση στη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και όχι στην ανάπτυξη περιβαλλοντοκτόνων μονάδων παραγωγής ενέργειας από ουράνιο και άνθρακα. βέβαια ελπίζω όσοι σκέφτονται την ενίσχυση με νέε κατασκευέ του πυρηνικού λόμπι να πήραν ένα μάθημα από την πρόσφατη συμφωνία τη τουρκία με τη ρωσία για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο άκου μια σεισμογενή όπου το αντιπυρηνικό κίνημα έχει αποτρέψει την κατασκευή του. Ε, Κύριε Τρεμόπουλε, χρονικό η ε, κυρία Μπαρμπανόβα έχει σηκώσει την ε, γαλάζια κάρτα τη. Συνεπώ, κύριε Τρεμόπουλε, ε, θα μπορούσε να σα κάνει μια ερώτηση. Θέλω Κυρία Παρβανόβα, με μεγάλη συντομία να ακούσουμε την ερώτησή σα. πρόεδρε, η κυρία Βαλεάν ε, είπε ότι οι Βουλγαροί δεν χρησιμοποίησαν σωστά τα κονδύλια τα οποία τους έχουν, ε, τα οποία έχει λάβει. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ο Μιλήτρια. Θα, Συγγνώμη, οι διαδικασίε είναι διαφορετικέ. Κύριε Παπανόβα, ε, παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σα, Η διαδικασία προβλέπει ερώτηση στον ομιλητή, όχι στην Κομισιόν. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε ερώτηση προ τον Επίτροπο. συνεπώ απορρίπτεται αυτή η ερώτηση και συνεπώ δεν θα σα απαντηθεί κιόλα. Για ένα λεπτό, ο λόγο στον κύριο Φανόρδεν. Ε, εκ των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πολέμησα για να εμποδίσω τον την πρόορη αποξήλωση του Κοσλόντουι. Ε, δεν ήταν αναγκαίο να, να κλείσουμε τις αντιδραστήρες για λόγους ασφάλειας τόσα χρόνια νωρίτερα. Το αποτέλεσμα, όπως προβλεπόταν, ήταν ε, να χρησιμοποιούμε ε, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη που είναι εντελώς ε, αντίθετη από περιβαλλοντικής πλευράς προς όλα τα πρότυπα και που προκαλούν μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά. Και τώρα προσπαθούμε ε, εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διορθώσουμε αυτή τη ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν δίκαιο είναι να αντιμετωπίσουμε τη Βουλγαρία όπω ακριβώ και άλλε χώρε που χρειάστηκε να κλείσουν ε, πρόωρα τι ε, και γυρέ ε, πυρηνικέ του εγκαταστάσει. Το αναγνωρίζει αυτό η Κομισιόν. Φυσικά ε, δόθηκαν πολλά χρήματα για αυτή την ε, αποξήλωση και παροπλισμό. Ε, Βεβαίω αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να ξοδευτούν αποτελεσματικά και ελπίζω η Κομισιόν να μα διαβεβαιώσει ότι θα το παρακολουθήσει. Επίση είναι σημαντικό να δούμε το θέμα τη της αποζημίωσης για την απώλεια της, του ενεργειακού δυναμικού της Βουλγαρίας. Θα πρέπει για να υπάρχει ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού ε, και επικοινομορφία στην ενέργεια η ε, Βουλγαρία να μπορεί να παράγει ενέργεια από άλλες πηγές. Ο κ. Φανόρταν, εκ μέρους της ΚΟΕ. Ευχαριστούμε μάλλον. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε τον κ. Φανόρταν. Ο κ. Ράνστορ. Εκ μέρους της ΚΟΕ. Το πρόγραμμα Κοσλοντούι δεν μπορεί να εστιαστεί μόνο στη χρηματοδότηση της μεταφοράς ραδιενεργών υλικών και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Βουλγαρία ταυτόχρονα με τη χρηματοδότηση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνεισφέρει και στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων. Διότι τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας, είναι από τα πιο ευάλωτα κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το είδαμε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το άρθρο 30 της ε, ε, συνθήκης προσχώρησης της ε, Βουλγαρίας δεν θα πρέπει να παραβιαστεί. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να διατηρεί τη συνέχεια με το άρθρο 30. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Τελειώνουμε αυτό το γύρο με την ε, παρέμβαση του κυρίου Στογιανόφ για δύο λεπτά εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε για ε, χρήματα που, και την αντιστάθμιση που θα δοθεί στη Βουλγαρία για το κλείσιμο του Κοσλοντούι που είναι και δίκαιη και έγκαιροι, Γιατί έχει εκτιμηθεί ότι υπάρχει απώλεια συνεχιζόμενη από το κλείσιμο των δύο μονάδων πολύ υψηλότερη από την αντιστάθμιση αποζημίωση που έλαβε. Γιατί φτάσαμε εδώ, όπως είπα και πριν, όπως και πριν, οι πιο ασφαλείς μονάδες στην Ευρώπη και αυτό το είπε ε, η Διεθνής Επιτροπή ατομικής ενέργειας, γιατί θα έπρεπε να κλείσει η ασφαλέστερη μονάδα και πώς έφτασε η έκθεση να πέσει στα χέρια των πρασίνων ε, που όπως ο Μάρκος Αντώνιος ε, ε, σκοπό είχαν το, το, το πώς θα γίνει η καταστροφή δεν θα πρέπει να είστε εσείς αυτοί που μας θα λέτε αυτά, γιατί η χώρα σας ε, έκανε εκβιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε πολύ περισσότερα λεφτά από τη Βουλγαρία. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τον Έλληνα συνάδελφο να σιωπήσει και να μην μας ε, λέει τι πρέπει να παίρνουμε και τι όχι. Οι πράσινοι ένα και μόνο στόχο είχαν. Είχαν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι με το κλείσιμο του Κοσλοντούι αυξήθηκαν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τώρα τολμούν να φερούν ε, κονδύλια από τη Βουλγαρία για να τα δώσουν αλλού, ε, για να σώσουν τα προσχήματα και να τα σώσουν απέναντι στους ε, εκλογείς που πώς είναι δυνατόν παρόλα τα μέτρα τους να αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, κάτι άλλο ε, που, στο οποίο έδωσε το παράδειγμα το Κόσλο Ντού ήταν υποδειγματικό. Το πώς οι παλιοί αντιδραστήρες μπορεί να συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά. Το μόνο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε στο μέλλον είναι αρνητικό μέσα από πολιτική ανοησία που οδήγησε σε κλείσιμο και εκαθάριση μιας σημαντικής ε, βιομηχανικής μονάδας. Ε, είσαστε πάρα πολύ κοντά στα όρια της αγένειας ε, ε, και σχεδόν έχετε ξεφύγει από τους κοινοβουλευτικούς ε, καλούς τρόπους. Δεν σας διακόψα από γενεοδορία. Η, η ομάδα των Πρασίνων δέχθηκε βαριά επίθεση και θέλω να σας αποδείξω ότι εμείς έχουμε την ικανότητα να ακούμε, πλην όμω, πρέπει να υπογραμμίσω ότι ήταν απρεπή η συμπεριφορά σα. Την επόμενη φορά θα σα διακόψω, δεν θα σα επιτρέψω να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο. Τελειώσαμε με τις παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων που ε, εξέφρασαν την γνώμη της ομάδας τους και περνάμε στις ε, τοποθετήσεις ξενόματος των ιδίων. Καταρχήν ο λόγος του κ. Στολογιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν, γιατί παρότι ανησυχούμε πολύ περισσότερο για την οικονομική κρίση από ότι οτιδήποτε άλλο, η Κομισιόν έχει το θάρρος να ασχολείται και με άλλα προβλήματα πέρα από τα οικονομικά. Και η Βουλγαρία νομίζω έχει το δικαίωμα να λάβει αυτά τα χρήματα τα οποία ε, της τα υποσχέθηκαν. Της τα υποσχέθηκαν για τον παροπλισμό αυτού του πυρηνικού εργοστασίου. Εγώ υποστηρίζω την ηλεκτρική ενέργεια ε, και θεωρώ ότι μπορεί να παράγεται με ασφαλή τρόπο από την πυρηνική ενέργεια. Και δεν νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους ε, που έχει θέσει σε ό,τι αφορά την πράσινη ενέργεια χωρίς την ε, κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων. Πιστεύω πραγματικά ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να χτίζει πυρηνικά εργοστάσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε μια συλλογική ευθύνη για αυτό το θέμα και θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τις ε, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρή και αυστηρή όταν αξιολογεί αυτά τα προγράμματα για την ε, οικοδόμηση νέων πυρηνικών εργοστασίων. Για δύο λεπτά ο κύριος Παλέκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και να υποστηρίξω το έγγραφο το οποίο συζητάμε. Επίσης, επίσης υποστηρίζω την ιδέα να δοθούν 300 εκατομμύρια είδη βοήθεια στη Βουλγαρία για την αποξήλωση των τεσσάρων μονάδων στο Κοσλοντούι μέσα σε μία τριετή περίοδο. Παράλληλα, η διαχείριση και ο έλεγχος των κονδυλίων αυτών θα πρέπει να γίνει με αυστηρό τρόπο. Θα πρέπει να σταματήσει η αδικία και να δείξουμε αλληλεγγύη όπως και στα άλλα κράτη-μέλη, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία που έλαβαν αντίστοιχη βοήθεια. Αυτές οι τέσσερις μονάδες ε, έχουν πάψει να λειτουργούν εδώ και αρκετό καιρό και επομένω είναι λογικό να κλείσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος και θα μας βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δεξιότητες και την εμπειρία των εργαζομένων στον σταθμό. Μετά το κλείσιμο το προσωπικό του σταθμού θα αντιμετωπίσει νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις. Με βάση την εμπειρία της Λιθουανίας μπορώ να σας πω ότι συνήθως ε, υπάρχουν απρόβλεπτα εμπόδια και τα χρονοδιαγράμματα γενικά δεν μπορούν να τηρηθούν. Γενικά συμφωνώ ότι η μερίδα του λέοντος ε, από τους πόρους θα πρέπει να πάνε στον παροπλισμό και στην αποθήκευση του πυρηνικού, των πυρηνικών αποβλήτων. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους που δούλεψαν. Νομίζω ότι η βουλγαρική κυβέρνηση με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς και τις κοινότητες ε, γύρω από το εργοστάσιο για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Είναι ε, πολύ, σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να λάβουν νέα προσόντα και νέες δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που έχουν και τις γνώσεις τους σε άλλες βιομηχανίες. Νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας θα πρέπει να δημιουργηθούν και νέες βιομηχανίες πιο φιλοπεριβαλλοντικές επίσης πρέπει να δημιουργηθούν. Ευχαριστώ κύριε Παλέκη. Παλέκης, ο κύριος Ζημάντσκι. Δεν έχετε σηκώσει το καρτελάκι σας, σας βλέπω όρθιο. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο παραπλησμός τεσσάρων μονάδων του Κοσλοντούι ε, προκάλεσε σημαντική μείωση της παραγόμενης ενέργειας και ασφαλώς έθεσε σε κίνδυνο την συνολική ασφάλεια τροφοδοσία στην ε, περιοχή και αύξησε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι προτείνουν να, να αμελήσουμε το πρόβλημα της ενεργειακή τροφοδοσίας. Όμως, ε, η αρχή της ελληνική ε, θα πρέπει να περτανεύσει. Δεν είναι δυνατόν η πυρηνική ενέργεια να υφίσταται αρνητικές διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο λόγος στην κυρία Κρέτκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόβλημα του παραπλησμού και της αποξύλωσης δεν είναι μόνο σημαντικό για το πώς θα λύσει η Βουλγαρία το πρόβλημα, αλλά η διαδικασία παροπλισμού επηρεάζει και τις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να υπάρξει παράδειγμα εδώ για την αντιμετώπιση πυρηνικών εργοστασίων. Το Κοσλοντούι πάντοτε απασχολούσε τους Ρουμάνους ιδιαίτερα μετά το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Γι' αυτό είναι σημαντικό η διαδικασία του παροπλισμού να συνοδεύεται και από μια δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης διότι ο κόσμος δικαιούται να ενημερώνεται και για τα, τις φάσεις που θα ακολουθηθούν και τους κινδύνους, τους τρόπους αντιμετώπισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Είναι σημαντικό αυτό. Για αυτό τα κονδύλια στη Βουλγαρία θα πρέπει να διακοπές. Φαίνεται να είναι επαρκή τα κονδύλια, αλλά είναι το εκτιμόμενο κόστος δεν υπάρχει προηγούμενο παροπλισμού στη Βουλγαρία. Ελπίζω να είναι αρκετά τα κονδύλια και προσεκτικός ο σχεδιασμός υπό την επιτήρηση όλων των φορέων ώστε το βουλγαρικό, η βουλγαρική αυτή περίπτωση να είναι παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Κρέτσο. Ο τελευταίος ομιλητής αυτή την σειρά, ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Οι χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προσχώρηση ανέλαβαν κάποιες σημαντικές οικονομικές και πολιτικές ε, δεσμεύσεις συμπεριλαμβανομένου του παροπλισμού των ατομικών εργοστασίων και την σωστή διάθεση των αποβλήτων ώστε να πληρούνται τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εργοστάσια ε, εφόσον δεν πληρούσαν τα πρότυπα θα έπρεπε να παροπλιστούν. Οι προϋποθέσεις σχετικά με τον παροπλισμό, την ασφάλεια των εργασιών παροπλισμού και οι πρόσθετες εργασίες προκάλεσαν και δημιούργησαν πρόσθετα εμπόδια για τις χώρες που δεν είχαν αρκετή χρηματοδότηση για την ε, διάθεση των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, απειλές για το περιβάλλον και άλλα προβλήματα. Συγχαίρω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει βοήθεια στη Βουλγαρία, γιατί χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Λιθουανία, η Βουλγαρία δεν θα μπορούσε να κλείσει σωστά τα εργοστάσια και να έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας. Τελειώσαμε το κατάλογο των ομιλητών. Κανένας δεν έχει ζητήσει την προσοχή του ματιού του Προέδρου. Συνεπώς ε, δεν έχουμε διαδικασία catch the eye. Περνάμε κατευθείαν στον Επίτροπο κ. Έτιγκερ, ο οποίος θα απαντήσει στις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Κύριε Έτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για την ε, ειλικρινή αντιπαράθεση σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν συνολικά συμφωνεί με την έκθεση αφού συμφωνεί και το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν να ενισχυθεί μέχρι το 2013 με 300 εκατομμύρια ευρώ η Βουλγαρία. Κατά τα άλλα, η έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των ασφαλών μέτρων αποξύλωσης και ότι υπάρχουν και ορισμένα προγράμματα στον ενεργειακό τομέα που θα πρέπει να ενισχυθούν. Τα κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν στοχευμένα. Είπατε και αυτό θα το παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Τις τροπολογίες σας τις λαμβάνουμε υπόψη. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη την ε, άποψη του Κοινοβουλίου ε, γιατί σε πολλά βελτιώνεται και ο κανονισμός. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ε, χρηματοδότηση της αποξύλωσης. Αυτό είναι ένδειξη αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Βουλγαρία. Η ασφάλεια κατά την αποξύλωση έχει την μέγιστη προτεραιότητα και αυτό το υπογραμμίζει η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και πάλι για την εργασία σας ε, και την συνάδελφο κυρία Χάρμς για την ε, έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Χάρμς έχει δύο λεπτά ως εισηγήτρια για την παρέμβασή της. Ευχαριστώ. Στο τέλος της συζήτησης θα ήθελα να σημειώσουμε ότι το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων στη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία έλαβε χώρα με βάση τη διεθνή πραγματογνωμοσύνη η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ήλεγξε τους αντιδραστήρες και είπε ότι με βελτίωση του εξοπλισμού είναι αδύνατο να τηρηθούν τα πρότυπα ασφαλείας όπως ίσχυαν στην παλιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή ήταν μια σοφή απόφαση και η απόφαση αυτή ε, δικαιώνει την αλληλέγγυα στάση μας με την αυριανή μας ε, στάση στην ψηφοφορία όπως στη Λιθουανία, όπως στη Σλοβακία και όπως στη Βουλγαρία θα πρέπει να ε, συμβάλλουμε στο κόστος του παροπλισμού. Δεύτερον, θα ήθελα άλλη μια φορά να πω ότι σε όλες αυτές τις χώρες, όπως και σε όλες τις ε, χώρες της Δυτικής Ευρώπης και διεθνώς, μέχρι τώρα καμία χώρα δεν ε, βρήκε ε, τέλεια λύση σχετικά με την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων. Έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια και εδώ και 30 χρόνια αναζητείται μια υπεύθυνη λύση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που, με την οποία πρέπει να ασχοληθούν κυρίως εκείνοι που τάσσονται υπέρ της τεχνολογίας, της πυρηνικής τεχνολογίας υψηλού κινδύνου. Γιατί η αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων θεωρώ και νομίζω ότι και η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρώπη συμπαρατάσσονται μαζί μου, είναι ανεπίλητος κίνδυνος ε, που από μόνος του συνηγορεί υπέρ της μη χρήσης της, πολιτικής, της πυρηνικής ενέργειας. Θα το συζητήσω και με τον κύριο Έτιγκερ και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάμστ. Έκλεισε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Αύριο το πρωί θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση από τις 10 έως τις 1 και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας, ε, για το χρόνο που διαθέσατε.